Hello everyone, if you want to take your seat. Καθίστε παρακαλώ να ξεκινήσουμε το τμήμα αυτό της συνεδρίασης που είναι κάπως ιδιαίτερο, κοινή συνεδρίαση με τους αδρούς μας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Μια πολύ σημαντική έκθεση συζητήσουμε. Την έκθεση για τη διπλωματία στον τομέα του κλίματος. Να καλωσορίσω όλους τους βουλευτές που ήρθαν εδώ σήμερα το απόγευμα Χαίρομαι που αποφάσισαν οι δύο επιτροπέ ε, ότι είναι σκόπιμο να ενώσουν τι δυνάμει του την έκθεση αυτή σε ένα σημαντικό θέμα όπω είναι αυτό τη διπλωματία στον τομέα του κλίματο. Και είναι και πολύ επίκαιρο θέμα εφόσον το Συμβούλιο ανέκρινε τα συμπεράσματά του πρόσφατα για το θέμα αυτό, 26 Φεβρουαρίου συγκεκριμένα. Και επειδή βέβαια είναι πραγματικότητα σήμερα η αλλαγή του κλίματος, επηρεάζει την ε, ζωή μας με πολύ απτό τρόπο. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε φιλόδοξοι και να επανεπιβεβαιώσουμε τις δεσμεύσεις μας για τη Συμφωνία των Παρισίων και του στόχου του, για να μειώσουμε τις επιπτώσεις του, της αλλαγής του κλίματος. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης να επανεπιβεβαιώσει τον ηγετικό της ρόλο στην κλιματική δράση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνηση που πρέπει να συμμετέχουν για τη διευκόλυνση του διαλόγου, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, συνεργασία μεταξύ κρατικών και μη κρατικών φορέων. Σε όλους αυτούς τους τομείς ε, η προσέγγιση μας ήταν πάρα πολύ επικοδομητική. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της αλυσίδας τροφίμων και η κλιματική διάσταση και στην εξωτερική πολιτική. Και αυτά είναι προφανή και για αυτούς τους λόγους είναι σημαντικό να συνεργαστούν οι επιτροποί μας για το θέμα αυτό και είμαι βεβαία ότι θα είναι ομαλή συνεργασία μα για να εκπέμψουμε ένα χειρομήνου. Προσβλέπω με ανυπομονησία τη συζήτηση για το σχέδιο έκθεση, συζήτηση που θα γίνει σήμερα. Και θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Κλάουσου Μπουχνέρ που αντικαθιστά τον κύριο Μακάλιστερ, πρόεδρο τη ΑΦΕΤ, σήμερα. να παρακαλώ λοιπόν να κάνετε τι αγωγικέ του Κύριε Μπουχνέρ, καλώ ορίσατε και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βαλεάν για την πολύ ευγενική σα αυτή εισαγωγή. Η έκθεση αυτή δεν είναι μόνο επίκαιρη, αλλά και πολύ σημαντική για εμάς. Μπορώ να μιλήσω για την δική μου εμπειρία σε πολλές αντιπροσωπείες. Το θέμα αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Νομίζω ότι με την έκθεση αυτή έχουμε μια πολύ καλή προσέγγιση που μπορούμε να υιοθετήσουμε. Πρώτον λέγεται ότι πρέπει να υιοθετήσουμε, μάλλον να εντοπίσουμε τις βασικές μας προτεραιότητες. Και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε σε όλες τις αντιπροσωπείες. Ήταν μεγάλο πλεονέκτημα κατά που αποφασίσαμε να συντάξουμε την έκθεση αυτή, αλλά δεν θα πω άλλα, δεν θα πω κάτι ακόμη, θα σταματήσω και θα δώσω το λόγο στην κυρία Ντάλη. Um, Ευχαριστώ και τους δυο σας. Εγώ σήμερα μιλάω εκ μέρους του Λάινεν, που είναι εισηγητής ε, για την διπλωματία στον τομέα του κλίματος. Δυστυχώς όμως δεν μπορούσε να είναι σήμερα παρόν. Μου ζήτησε λοιπόν να εκφράσω τις ευχαριστίες του στον Αρνελή, στον συνεισηγητή, για την πολύ επικοδομητική συνεργασία που είχαν τους τελευταίους μήνες. Ο Γιώ Λάινεν θέλει να ακούσει και τις απόψεις των άλλων σκιωδών εισηγητών, αλλά και τις απόψεις της Κομισιόν για το σχέδιο έκθεσης. Η έκθεση αυτή του Κοινοβουλίου είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να βελτιώσουμε τι σοβαρέ δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει για την κλιματική δράση και θα συνεισφέρει η έκθεση και στη εφαρμογή τη Συμφωνία του Παρισιού και στην Ένωση και παγκοσμίω. Πρώτη φορά ασχολείται το Κοινοβούλιο ιδιαίτερα με την κλιματική διπλωματία και είναι και μια ευκαιρία για μας να συνεισφέρουμε πριν και την COP14 και το διάλογο Ταλανό θα λάβει χώρα Είναι πάρα πολύ θετικό να γίνει αυτό και να είναι μια κοινή προσπάθεια μεταξύ των Επιτροπών ΑΦΕΤ και ΕΝΒΙ, γιατί η κλιματική διπλωματία χρησιμοποιεί μέτρα τη εξωτερική δράση και μέσα τη εξωτερική δράση για την κλιματική προστασία. Το σχέδιο έκθεση ήδη διατυπώνει συστάσει προ την Κομισιόν και την ΕΙΕΔ, αλλά και τα κράτη-μέλη. Με στόχο μια πιο στρατηγική, συνεκτική διπλωματία από πλευρά Ένωση για στον τομέα του κλίματο, που θα επηρεάζει. Τρει προτεραιότητε θέλω να αναφέρω. Αν είναι, θέλουμε να είναι επιτυχημένοι, η πολιτική θα πρέπει να έχει την απαιτούμενη φροδοξία του απαιτούμενου πόρου και τι απαιτούμενε στρατικέ συνεργασίε και φαντάζομαι ότι σε αυτά θα προσθέσει ε, τη δική του άποψη και ο Αρνελίτς ο συνεισηγητή. Μπαίνουμε σε μια κρίσιμη φάση της υλοποίηση συμφωνία των Παρισίων. Την ειδική έκθεση του IPCC την περιμένουμε για, τον, για το φθινόπωρο του 2018. Και έτσι θα έρθουμε αντιμέτωποι με την ανάγκη να μειώσουμε την υπερθέρμανση του κλίματος 1,5 βαθμό Κελσίου. Στιγμή αλήθεια για την παγκόσμια κοινότητα. Έχουμε τον πρώτο διάλογο Ταλανό και ελπίζουμε και το book ε, να έχει υλοποιηθεί μέχρι τότε. Να δούμε λοιπόν πόσο στεναρή θα είναι η υλοποίηση της συμφωνίας. Και να δούμε και αν θα τηρηθούν υποσχέσεις που έχουν αναλυφθεί. Ο Διόλαβο Ταλανό απαιτεί από όλες τις ε, πλευρές ε, να παρουσιάσουν τη συνεισφορά τους για μια κοινωνία με μηδενικέ εκπομπέ, κλιματική αλλαγή. Ήδη υποβαθμίζει τη, το συνθήκε διαβίωση. Αυξάνει ξηρασίε, πλημμύρε, Είχαμε το ε, διάσκεψη του κλίματος για το κλίμα πέρυσι, που δείχνει πόσο απειλεί το περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, πόσο απειλεί τη σταθερότητα και την ειρήνη στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο. Στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει την πολιτική και οικονομική ικανότητα να είναι ηγέτης στον τομέα της κλιματικής δράσης. Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, χρειαζόμαστε στρατηγικές εταιρικές σχέσεις. Όχι μόνο να είμαστε δραστήριοι διαμεσολαβητές στο πλαίσιο των Εθνών και των σχετικών διαπραγματεύσεων, αλλά και ε, απέναντι σε οργανώσεις όπως είναι ο Διεθνής Οργανισμός ή η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας. Με μεγαλύτερο επαγγελματισμό, να ακολουθούμε μια στρατηγική συγκεκριμένη, να αξιοποιούμε τους πόρους μας, ε, τα μέσα μας και να αντιμετωπίσουμε διάφορα επίπεδα και να έρθουμε σε επαφή με διάφορους παράγοντες με στοχευμένο τρόπο. Στην COP24 ε, θα πρέπει να αναβιωθεί η συμμαχία των κρατών. Θα πρέπει να συνεργαστούμε επίσης με τις περιφερειακές αρχές, με τις εταιρείε, τους ΜΚΟ και θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τις αναδυόμενες οικονομίες. διαφορετικές οικονομίες, διαφορετικά πολιτικά συστήματα πρέπει να συνδυαστούν, όμω. είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Και η σχέση με την Κίνα είναι κάτι πολύ σημαντικό για την κλιματική δράση. Θέλουμε στενή συμμαχία πριν την COP24 και μετά όμως από αυτή Μία συμμαχία με την Κίνα μπορεί να εμβαθυνθεί η συνεργασία σε διάφορους τομείς, όπως ανέσουμε πηγές ενέργειας και η ηλεκτροκίνηση. Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης θα πρέπει να αγηθεί της διαδικασίας ανάπτυξης του αγο... της ε, αγοράς άνθρακα με το σύστημα ETS και σε σχέση με την Κίνα και με άλλες αγορές όπως είπα και Καναδά. Θα πρέπει να ξεπεράσει την πολιτική διπλωματία, η κλιματική διπλωματία να περιλαμβάνει από την επιστήμη, από τις επιχειρήσεις, Και θα πρέπει να υπάρξουν και στρατηγικές εξαγωγών. Να χρησιμοποιήσουμε τη γνωσή μας και την ε, ηγετική μας θέση για τη δημιουργία υποδομών και δυνατοτήτων σε άλλες χώρες. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να γίνει ένας διπλωματικός εταίρος και να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητε του και τις αρμοδιότητες εκχωρώντας τις και σε τρίτους με πιο αποτελεσματικό τρόπο στόχος να έχουμε μια νέα στρατηγική για τη διπλωματία στον τομέα του κλίματος. να γίνουμε κινητήριος μοχλός για την κλιματική δράση σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της κλιματικής διπλωματίας. Στο ό,τι αφορά απαιτούμενους πόρους. Μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο μπορεί να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Πρέπει να έχουμε λοιπόν την παγκόσμια υποστήριξη. Στην COP24 πρέπει να στείλουμε μηνύματα σαφή και διαφυσβήτητα. Μπορεί να είναι ένα ισχυρό όπλο αυτή η κλιματική διπλωματία για να πετύχουμε από άλλες ανεπτυγμένες χώρες μεγαλύτερη δέσμευση. Για να είναι αποτελεσματική η κλιματική διπλωματία και να προωθήσει το θεματολόγιο το κλιματικό θα πρέπει να έχει του απαιτούμενου πόρου Το σχέδιο έκθεση, προτείνει να αξιολογηθεί και η χρηματοδότηση και το ανθρώπινο δυναμικό για να κλείσουν κάποια κενά που υπάρχουν στον τομέα των δυνατοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό πρέπει να αντικατοπτριστεί και στο πολιτές πλαίσιο σημαντικό στόχο κατά του ΠΔΠ. Υπάρχουν δημοσιονομικέ πιέσει, αλλά πρέπει να διατεθούν επαρκή πόροι για το κλίμα. Όχι απλά αυτοί που έχουν ήδη διατεθεί στο τρέχον πλαίσιο, αλλά να αυξηθούν. Εμεί ζητάμε 30% και θα το επαναλάβουμε και στην έκθεση αυτή αυτό το αίτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την ήπια δύναμη αλλά και την κρηματοοικονομική ε, της δύναμη κάποια άλλα σημεία που θέλει να αναφέρει ο είναι και αναφέρονται και στην έκθεση είναι ότι είναι κατεπίγουσα ανάγκη για ανάληψη δράση. Δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε βέβαια το επίπεδο φιλοδοξία, όμω αναμφίβολα πρέπει να είναι πάνω από τους στόχους του 2030 που ορίσαμε το 2014 πριν τη σύναψη της συμφωνία των Παρισίων. Δεν είναι τι έχει να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τι πρέπει να προσφέρει. Αυτό είναι το θέμα χωρίς και την έκθεση του IPCC και χωρίς το διάλογο τάλανο, ξέρουμε ότι η μείωση του 40% δεν θα μας βάλει στο σωστό δρόμο για την εξάλληψη των εκπομπών μέχρι τα μέσα του αιώνα. Η Ευρώπη που είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο δεν μπορεί να ε, αποποιηθεί των ευθυνών της. Και θέλουμε να στήσουμε στην έκθεσή μας από Κομισιόν και κράτη-μέλη να είναι έτοιμα να υλοποιήσουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη αξιοπιστία. Άρα πρέπει να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στο διάλογο του Θέλουμε μετριασμό ε, της κλιματικής αλλαγής και αύξηση των χρηματοοικονομικών εισφορών από τα άλλα κράτη. Αυτό για να το πετύχουμε πρέπει και εμείς να προσφέρουμε κάτι των προτέρων. Πρέπει να αναπτύξουμε μια στρατηγική ενωσιακή για το 2050. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας του Παρισιού ένα νέο σχέδιο για το 2050 με μέτρα συγκεκριμένα για το μετριασμό τη αλλαγή του κλίματος. Αυτό θα βοηθήσει και στο εσωτερικό επίπεδο να γίνει κατανοητό τι βήματα πρέπει να γίνουν το 2020 και το 2030. Ήδη είμαστε παράδειγμα για άλλε ε, περιφέρειες και υπήρου. Κλιματική δράση δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα σε αντιδιαστολή με την ανάπτυξη τα υψηλά πρότυπα. Αυτό το έχουμε αποδείξει. Η Συμπερασματικά τώρα είναι μια νέα έννοια αυτή η διπλωματία στον τομέα του κλίματο, αλλά νομίζω ότι εμεί πρέπει στο Κοινοβουλίο να στείλουμε το μήνυμα ότι στηρίζουμε την αυξαμένη διπλωματία στον τομέα του κλίματο θέλουμε να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή. Το σχέδιο έκθεση είναι περιορισμένο ε, στους χαρακτήρες. Ε, θα προσπαθήσει λοιπόν ο Γιώ ε, να δώσει και άλλες συγκεκριμένες προτάσεις που θα καταστήσουν πιο σαφή αυτή την πρόταση. Τώρα θα πάρει το λόγο κύριος Αρνελίτς. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία και κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που μπορούμε να κάνουμε σήμερα αυτή τη συζήτηση σε σχέση με τα επιτεύγματα μέχρι στιγμής. Πραγματικά η έκθεση αυτή έρχεται την κατάλληλη στιγμή καθότι βλέπουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε αποχωρούν από τη Συμφωνία των Παρισίων. Και όπω είπατε και εσεί, κύριε Πρόεδρε, η κλιματική αλλαγή αποτελεί πραγματικότητα. Δεν το πιστεύουν αυτό όλοι, όπω ο κύριο Τράμπα. Αλλά έχουμε και κάποιε. Ε, ακροδεξιές πολιτικές ομάδες, ακόμα και η EFD στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι πολιτική ομάδα από την Γερμανία, θεωρούν ότι δεν αποτελεί πραγματικότητα κλιματική αλλαγή. Αυτό προφανώς δεν αληθεύει. Θα πρέπει λοιπόν από κοινού να δείξουμε μια ενωμένη στάση. Το Συμβούλιο επίσης έχει ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό της διπλωματίας στον τομέα του κλίματος, προχωρώντας συμπεράσματα ήδη το Φεβρουάριο και η Επιτροπή των Περιφερών επίση είχε ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό και κατέληξαν σε ένα σχέδιο γνωμοδότησης από την Επιτροπή όσον αφορά το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και την ε, ενέργεια. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φορεί από διάφορα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ασχολούνται με το ζήτημα αυτό. Η ίδια η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει να εντάσσεται όλο και περισσότερο σε αυτό το οποίο ονομάζουμε διπλωματία στον τομέα του κλίματο, κυρίω μέσω τη εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνείς διασκέψεις όπως αυτή που έλαβε χώρα στο Μόναχο για την ασφάλεια έχει αναλυθεί και το ζήτημα αυτό της διπλωματίας στον τομέα του κλίματος. Για πρώτη φορά η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ασχολείται πλέον με το ζήτημα αυτό για τους λόγους αυτούς που έθεσε μέσω του συναδέλφου ο κύριος Γιολάινεν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί το στην κόψα, αλλά βλέπουμε τώρα ότι θα πρέπει να προσεγγίσουμε περισσότερο όλες τις χώρες του πλανήτη προκειμένου να εφαρμοστεί πλέον η Συμφωνία των Παρισίων και το ψήφισμα των Παρισίων. Και πάλι θα πρέπει στον τομέα της διπλωματίας μαζί με όλου του εμπλεκόμενου παράγοντε στο τομέα του περιβάλλοντος να καταφέρουμε να κρατήσουμε σε υψηλό επίπεδο και ω βασική προτεραιότητα την Συμφωνία των Παρισίων. Τρει πυλώνε έχουμε. Καταρχά, θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποτελέσει σημαντικό το παράγοντα όσον αφορά τη διπλωματία στον τομέα του κλίματο. Δεύτερον, θέλουμε να ενσωματώσουμε τη διάσταση του κλίματος σε όλες τις εξωτερικές δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτον θέλουμε να έχουμε το απαραίτητο προσωπικό και την απαραίτητη χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου η δράση του στον τομέα του κλίματο να είναι πιο φιλόδοξη και πιο αξιόπιστη. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να αναλυφθούν απαραίτητε πρωτοβουλίε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση Έχουμε έπειτα την απαραίτητη ορολογία όσον αφορά του τι είναι η διπλωματία στον τομέα του κλίματο. Αποτελεί μια στοχευμένη εξωτερική πολιτική για την προώθηση τη πολιτική για την αντιμετώπιση του κλίματο προ τα έξω, προ τα έξω, προς άλλου παράγοντε. Ασχολούμεθα με συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Δημιουργούμε εταιρικέ σχέσει με άλλε κυβερνήσει ή μη κυβερνητικού παράγοντε προκειμένου να μειώσουμε, να μετριάσουμε τι επιπτώσει τη κλιματική αλλαγή. Ποιες τώρα είναι οι βασικές μας προτεραιότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε ότι είναι από τους σημαντικότερου παράγοντες στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής συνέβαλε πάρα πολύ στο να συναυθεί η Συμφωνία των Παρισίων και να προωθηθεί ένα θεματολόγιο για τις κλιματικές αλλαγές. Προκειμένου όμως να καταφέρει να δραματίσει το το ρόλο τη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παραμείνει αξιόπιστο παράγοντα, να δείξει ηγετική στάση και να συμβάλλει όλο και περισσότερο στον τομέα τη διπλωματίας, στον τομέα του κλίματο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική για κοινέ ενωσιακέ προσπάθειες για τον τομέα του κλίματο και θα πρέπει να είναι συνεκτική στάση αυτή και να φέρνει μαζί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να καταφέρουμε να προωθήσουμε το ζήτημα του κλίματο στο θεματολόγιο εξωτερικών υποθέσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχει ένα σύστημα υποβολή εκθέσεων για την στρατηγική για το κλίμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταφέρουμε να εμπλέξουμε περισσότερο τι επιτροπέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα μπορούν να πηγαίνουν και σε άλλε χώρε. Ε, για παράδειγμα, κάθε φορά που τα αντιπροσωπείε προ τρίτε χώρε για το ζήτημα του κλίματο, θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχει και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Περιβάλλοντο. Θα πρέπει να καλλιεργήσουμε περισσότερε σχέσει για το ζήτημα του κλίματο με άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ από άλλα κοινοβούλια, καθώ επίση και με περιφερειακέ οργανώσει, όπω για παράδειγμα στην Αφρική ή στην περιοχή τη Καραϊβική και θα πρέπει επίσης να έχουμε και τον απαραίτητο προϋπολογισμό προκειμένου να έχουμε και μια φιλόδοξη δράση. Ήδη στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα του κλίματος, να έχουμε συγκεκριμένε γραμμές του προπολογισμού πλέον οριζόντιες, οι οποίες να ασχολούνται και να δίνουν κονδύλου ουσιαστικά στο ζήτημα της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Είναι πολύ σημαντικό να προωθηθεί η Ατζέντα 21, καθώς επίσης και η Συμφωνία των Παρισίων και θα πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο τη συμβολή μας όσον αφορά τους βιώσιμους στόχους, ε, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ένας από τους στόχους αυτούς είναι και η κλιματική αλλαγή και θα πρέπει του χρόνου στη συνεδρίαση που θα γίνει στη Νέα Υόρκη να έχουμε πλέον να από απτά αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μία συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία θα δώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα μας δοθεί και η δυνατότητα και σε εμά να εργαστούμε για την επίτευξη αυτού του στόχου. Θέλουμε λοιπόν μια συντονισμένη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και μια σφαιρική πολιτική για την κλιματική διπλωματία. Χρειαζόμαστε επίσης μια ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά, μιας, όσον αφορά τη διπλωματία στον τομέα του κλίματος. Θέλουμε σε αιτήσια βάση να υπάρχουν συστάσεις, καθώς επίσης και συντονισμένη δράση για την κλιματική αλλαγή. Ζητούμε επίσης να γίνει καλύτερη χρήση των αντιπροσωπιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς επίσης και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης κάθε φορά που πηγαίνουμε σε τρίτες χώρες. Ξέρετε ότι ε, ήδη στις αντιπροσωπείς Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ηνωμένε Πολιτείε, καθώς επίσης και σε άλλες χώρες, έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το ζήτημα αυτό της προώθησης της πολιτικής μας για την κλιματική αλλαγή. Ξέρετε ότι ήδη υπάρχει ο συντονισμός αυτός μεταξύ κρατών μελών. Κάθε μήνα, για παράδειγμα, υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των αντιπροσωπιών των κρατών μελών και υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια για αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνεται από ενωσιακής πλευράς όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Ξέρετε ότι Στι Ηνωμένε Πολιτείε ήδη υπάρχει μία επαφή με τα απαραίτητα θεσμικά όργανα, το Λευκό Οίκο αλλά και άλλα, προκειμένου να μπορούμε να προωθούμε περισσότερο μία ενιαία στάση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό να εμπλέκονται περισσότερο και γενικέ διευθύνσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γενικά να έχουμε ένα ενιαίο μέτωπο. Επίση, χρειαζόμαστε μία στενή συνεργασία με τοπικούς, με, με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, με το τοπικό λεγόμενο επίπεδο, καλύτερη συνεργασία όσον αφορά και την προώθηση της πολιτικής μας για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, αλλά και για την προώθηση τοπικών οικονομιών με χαμηλότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ξέρετε ότι ε, ήδη πριν από λίγο καιρό έγινε μια σημαντική συνδιάσκεψη και με τις χώρες γειτονίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες παράγουν ορυκτά καύσιμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και συνήθως το πολλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι το ζήτημα των κλιματικών αλλαγών επηρεάζει πάρα πολύ και τη μετανάστευση και την προσφυγική κρίση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε λοιπόν μια πιο ενισχυμένη συνεργασία με τρίτες χώρες για τον τομέα της ενέργειας και ιδιότερα για τις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε περισσότερο με αναπτυσσόμενες και αναβιώμενες χώρες, καθώς επίσης και με επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών, καθώς επίσης και με την επιστημονική κοινότητα. Σαφώς λοιπόν ε, έχουμε αποκομίσει ήδη από τις τελευταίες εβδομάδες μια πολύ επικοδομητική ε, εμπειρία. Έχουμε συντάξει πλέον το σχέδιο αυτό έκθεσης. Είναι σημαντικό να καταφέρουμε να προσεγγίσουμε και χώρες όπως το Ιράν που έχουν αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα και στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά τις πολυμερείς εξωτερικές σχέσεις. Είναι σημαντικό να καταφέρουμε λοιπόν να εμπλέξουμε και χώρες εν μέρη απομονωμένες όπως το Ιράν, ανοίγοντά τους την πόρτα στη διπλωματία στον τομέα του κλίματος. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να τονίσουμε και την πτυχή της ασφάλειας όσον αφορά τι κλιματικέ αλλαγέ. Ενδεχομένω η πτυχή αυτή τη ασφάλεια να ευαισθητοποιήσει τι ΗΠΑ ή τον πρόεδρο Τραμπ, προκειμένου να συνεργαστεί περισσότερο μαζί μα εν τέλει και για το ζήτημα τη κλιματική αλλαγή. Νομίζω πάντω ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει σαφώ να το κρατήσουμε επιτάπητο στι επαφέ που έχουμε με την Αμερική. Προσβλέπουμε στι τροπολογίε που θα υποβάλλετε προκειμένου να βελτιωθεί το σχέδιο αυτό έκθεση που έχουμε υποβάλει προσβλέπουμε στις παρατηρήσεις των σχεδόν εισηγητών και των υπόλοιπων συναδέλφων από την Επιτροπή, από τις δύο Επιτροπές μάλλον, να ευχαριστήσω και τις γραμματείες των δύο Επιτροπών μας, οι οποίες συνέβαλαν πάρα πολύ στο να φτάσουμε, στο, στο σημείο που είμαστε σήμερα. Και να ευχαριστήσω και τους συνάδελφους και από τις δύο Επιτροπές, οι οποίοι συνεισέφεραν πάρα πολύ στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Πρόεδρος. Καλούνται οι σκιώδεις ηγητές να πάρουν τώρα το λόγο και να υποβάλουν παρατηρήσεις ή ερωτήσεις σε αυτή την κοινή έκθεση. Δύο λεπτά θα έχει το καθένας. Έχουμε μόνο έναν εισηγητή από την ΑΦΕΤ και την ΕΝΒΗ. Ενδεχομένως να μπορέσετε να μιλήσετε λοιπόν και τέσσερα λεπτά, αντικαθιστώντας έτσι και τον συνάδελφο της άλλης επιτροπής. Ο κύριος Πέτερλε είναι εδώ. Πολύ ωραίο. Θα μπορείτε να μιλήσετε και εξ ονόματος Ιδίας Σουίτσα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η κυρία Σουίτσα. Εκ μέρους ε, της κυρίας Σουίτσα, αγαπητοί συνάδελφοι, σας συγχαίρω για την εξαιρετική έκθεση. Η κλιματική αλλαγή απειλεί τη σταθερότητα, την ειρήνη και επηρεάζει σημαντικά πολλές ε, ε, διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής. Γι' αυτό το λόγο η κλιματική αλλαγή μπορεί να συμβάλλει στην εξωτερική πολιτική, σε στρατηγικές συνεργασίες και συνεργασίες με διάφορους παράγοντες ε, και εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα και ξεπερνώντας έτσι του, ε, τα συνηθισμένα όρια της κλιματικής ε, ε, πολιτικής. Προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας, η, κλιματική αλλαγή, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να γίνει στρατηγικός στόχος και να εντάξουμε την κλιματική αλλαγή στα αναπτυξιακά προγράμματα και σε όλες τις εξωτερικές δράσεις. Η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία των Παρισίων θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ευκαιρία να ηγηθεί τις δράσεις για την καταμολέμηση της κλιματικής αλλαγής και υποστηριχτούν οι στόχοι μας. Και αυτό θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε. Ο υπόλοιπο κόσμο μπορεί να βασιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να υλοποιηθεί μια φιλόδοξη κλιματική πολιτική πρέπει να συνεργαστούμε με τις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες και να βασιστούμε, βασίσουμε όλες τις προσπάθειές μας στη κλιματική διπλωματία. Αυτά έγραψε ο κύριος Ντούβρο Καρσουίτσερ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα εκ μέρους του ε, κυρίου Σμέρτσελη θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές για αυτή την εξαιρετική και ισορροπημένη έκθεση για ένα πολύ σημαντικό ε, ζήτημα. Η ε, έκθεση αυτή επιμένει στο στρατηγικό χαρακτήρα της ε, κλιματικής δράσης, η οποία πρέπει να ενταχθεί και στην εξωτερική μας πολιτική. Η έκθεση επαναβεβαιώνει τις δεσμεύσεις των ε, ως προς τους στόχους της ε, Συμφωνίας των Παρισίων μετά την αποχώρηση των ΥΠΑ ε, από την Συμφωνία. Είναι απαραίτητη μια ενοποιημένη δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας. Οι στρατηγικές συνεργασίες με διάφορους φορείς είναι πρωταρχικής σημασίας και αυτό θα ενθαρρύνει τους διάφορους παράγοντες να εμπλακούν στις απαραίτητες δράσεις. Και είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε τα υφιστάμενα εργαλεία, ωστόσο δεν έχουμε τα απαραίτητα μέσα για να υλοποιήσουμε τη στρατηγική μας. Η έκθεση αυτή εστίασε στη γενικότερα θέματα και όχι σε λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι ήταν μια υγιής προσέγγιση. και καλό θα ήταν αυτή η έκθεση να ενταχθεί σε όλα τα προγράμματα δράσης. Είναι σημαντικό να εστιάσουμε στα θέματα της ασφάλειας, του νερού, των τροφίμων, μιας και πρόκειται για πολύ σημαντικά προβλήματα που μπορούν να ενταθούν στο μέλλον. Ήταν τιμή μου που είχα τέσσερα λεπτά στη διάθεσή μου για να ε, εκφράσω τις παρατηρήσεις μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ και στους δύο κυρία Πέταλη και κύριο Σουίτσερ και εκ μέρους του ECR, κανείς, εκ μέρους την, της Άλντε, που θα μιλήσει εκ μέρους του κυρίου Πάιτ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές για την ισορροπημένη και φιλόδοξη αυτή έκθεση. Και θα ήθελα να τονίσω ότι όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή και όχι τα μονομένα κράτη-μέλη που θα πρέπει να προωθήσουν το ζήτημα της διπλωματίας στον τομέα του κλίματος και να δώσουν το παράδειγμα στον αφορά το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίω στα πλαίσια των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή να προωθήσουμε περισσότερο στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση το ζήτημα τη κλιματική αλλαγή. Οι αντιπροσωπείε τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πλέον να έχουν και προσωπικό πιο εξειδικευμένο στο ζήτημα τη κλιματική αλλαγή. Δύο συγκεκριμένε παρατηρήσει τώρα. Πρώτον, συμφωνώ ότι θα πρέπει να τεθούν θεματικέ προτεραιότητε συνεργασία στο ζήτημα της διπλωματία στον τομέα του κλίματο. Μια τέτοια θεματική προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η μελλοντική διπλωματία στον τομέα του κλίματος, ιδίως στον τομέα της, στην περιοχή της Αρκτικής. Θα πρέπει εδώ πέρα να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση στην Αρκτική και το γεγονός ότι έχουμε το πολύ σημαντικό φαινόμενο της τήξης των πάγων. Πρώτον λοιπόν αυτό. Δεύτερον, επαφή με την κοινωνία των πολιτών και με τους μη κυβερνητικού οργανισμούς. Αυτό αναφέρθηκε ήδη από τους συνεισηγητές και μνήα γίνεται στο σχέδιο έκθεσης. Θα ήθελα λίγο εδώ πέρα να επεκταθούμε περισσότερο. Συμφωνώ με τα όσα λέγονται στην έκθεση και επιπλέον πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να ενισχύσουμε περισσότερο τη θέση της γυναίκας, ιδίως όσον αφορά την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη και αυτό μπορεί να συμβάλλει περισσότερο σε μια πιο φιλοπεριβαλλοντική στάση που θα μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής ε, αλλαγής. Τώρα να μιλήσω εξ ονόματος του ε, συναδέλφου που απουσιάζει. Θεωρεί και αυτός ότι το κείμενο είναι καλό, θεωρεί ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Υπάρχουν ένα-δυο ζητήματα που, τα οποία θα θέλει να προσθέσει στην έκθεση αυτή. Πρώτον, λέει ο συνάδελφος ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή συνδέεται και με το φαινόμενο της μετανάστευσης. Δεύτερον, θα πρέπει επίσης να αναφέρεται στην έκθεση ότι οι επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής είναι πιο έντονες στην περιοχή της Τρακτικής, περισσότερο από οπουδήποτε αλλού. Και τρίτον, ο συνάδελφος θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο ζήτημα τη συμπεριφορά του κυρίου Τραμπ, ο οποίο αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Συμφωνία των Παρισίων και θα πρέπει να γίνεται επίση και μια αναφορά στο ότι περιμένουμε ακόμα η Ρωσία και αυτή με τη σειρά τη να επικυρώσει τη Συμφωνία των Παρισίων. Αυτά είχα να σα πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιατεμάκη, σα ευχαριστούμε, λέει πρόεδρο. Οι πράσινοι τώρα έχουν τον λόγο. Ο κύριο Αφρόντε. Θα μιλήσετε και τον κύριο Νταλούντε. Έχετε το λόγο σε κάθε περίπτωση πάντως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα-δύο σημεία να θίξω κι εγώ, κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ ότι ε, το σχέδιο έκθεση είναι ήδη αρκετά πλήρε και ήδη από τι ε, παρουσιάσει που γίνονται σήμερα από του δύο συγητέ φαίνεται ότι ε, ασχολούνται με πολλά διαφορετικά ζητήματα αλλά και σε βάθο, όχι μόνο επιφανειακά. Του των λεχθέντων υπάρχουν κάποια σημεία που θεωρούμε ότι πρέπει να τονίσουμε λίγο περισσότερο. Ένα από αυτά, κατά την άποψή μα, είναι το ότι θα πρέπει να προτείνουμε ακόμα πιο δυναμικά την ανάληψη δράσης, ιδίως όσον αφορά την πρόληψη, την ασφάλεια, την ασφάλεια των υδάτων, την ποιότητα του αέρα και ότι θα πρέπει να, αναφερθούμε επίσης και στην περιοχή νότια της Σαχάρας, περιοχές δηλαδή όπου έχουμε σημαντικά φαινόμενα λειψιδρίας, έλλειψη βασικών τροφίμων τα οποία αποτελούν βέβαια επιπτώσεις έντοπλων συγκρούσεων που έχουν πλήξει την περιοχή αυτή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε λοιπόν για κοινωνική ανισότητα, μετανάστευση, φτώχεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν σε επίπεδο διπλωματίας και εφόσον μιλάμε και διπλωματία στον τομέα του κλίματος να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτή την περιοχή. Το ίδιο το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του κάνει μια σχετική αναφορά στην υποσαχάρη αυτή περιοχή. Παράλληλα, θεωρούμε ότι ένα ακόμα σημείο το οποίο θα πρέπει να θίγουμε λίγο περισσότερο, σε ορισμένου μπορεί να φαίνεται λίγο δευτερεύον, είναι η ίδια η ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών. Ήδη από τη Eurostat γνωρίζουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε είναι ενήμεροι για την κλιματική αλλαγή, τα ποσοστά εδώ είναι πολύ θετικά, αλλά κατά την άποψή μα δεν υπάρχει η απαραίτητη ενημέρωση όσον αφορά τη διασύνδεση ανάμεσα σε κλιματικές αλλαγές και μετανάστευση, ένδια και γενικότερα μετατόπιση των πληθυσμών. Θεωρώ ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε θα πρέπει να γνωρίζουν περισσότερο ότι τα φαινόμενα αυτά είναι αλληλένδετα και ότι αντιμετωπίζοντα την κλιματική αλλαγή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και την προσφυγική κρίση. Είναι σημαντικό λοιπόν μια σχετική αναφορά να γίνεται και στην έκθεση, προκειμένου να υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική δράση για το μετριασμό τη κλιματική αλλαγή, με απότερο στόχο όμω την αντιμετώπιση άλλων αρνητικών φαινομένων, από πλευρά Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων έχουμε ήδη ετοιμάσει κάποιε τροπολογίε ορισμένες εκ των οποίων έχουν ε, ως στόχο να τονίσουν το ρόλο που μπορεί να δραματίσει η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής προκειμένου να προλάβουμε μελλοντικές συγκρούσεις θα υποβάλουμε βέβαια και κάποιες άλλες τροπολογίες λίγο πιο συγκεκριμένες σε ένα μεταγενέστερο στάδιο. Θεωρώ πάντως ότι η εργασία που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμή είναι εξαιρετική και υπάρχει απλώς ένα μικρό περιθώριο βελτίωσης, θεωρώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει γκουε τώρα. Θα μιλήσετε και την κυρία Τέρες Μαρτίνες. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Uh, Είμαστε υπέρ τη uh, έκθεση αυτή, uh, λέει ο κύριο Κούλογλου. Υποστηρίζουμε τις πτυχέ πτυχές έκθεση αυτή Να θίξω πολύ γρήγορα κάποια ζητήματα. Η διπλωματία στον τομέα του κλίματο στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι αξιόπιστη αν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τι δεσμεύσει στα πλαίσια τη Συμφωνία των Παρισίων. Θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού στα πλαίσια του φυστάμενου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Τρίτον, θεωρούμε ότι όντω είναι πάρα πολύ σημαντικό η διάσταση τη διπλωματία στον τομέα του κλίματο να ενταχθεί στι συμφωνίε εμπορίου και επενδύσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος εξορθολογισμό των προγραμμάτων αυτών προκειμένου τελικά να γίνεται και πιο αποτελεσματική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, είναι σημαντικό να μην υπάρχει διασύνδεση ανάμεσα στην απόσυρση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία των Παρισίων και το Brexit. Τα δύο αυτά ζητήματα δεν συνδέονται, θεωρούμε. Τώρα, η εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει τι απαραίτητε δυνατότητε προκειμένου να παρακολουθεί τι κλιματικέ αλλαγέ, να αξιολογεί του κινδύνου και να προχωρήσει απαραίτητε ενέργειε για την πρόληψη των συγκρούσεων και επίση να μπορεί να συνδέει περισσότερο τα φαινόμενα κλιματική αλλαγή με το ζήτημα των συγκρούσεων. Να ευχαριστήσω τους δύο συνεισηγητές και επιφυλασσόμεθα να υποβάλουμε και εμείς για το κείμενο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε συναδέλφους από το EFDD. Λοιπόν, τώρα μπορεί να πάρει οποιοδήποτε άλλο το λόγο. Ποιο θέλει να πάρει το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ. Ναι, ναι, απλώς ενημερώστε τη γραμματεία ώστε να σας, συμπεριλάβει στον κατάλογο αγορητών μόνο οι σκιώδει ναι. ε, εισηγητέ ήταν εγγεγραμμένοι μέχρι στιγμή. γι' αυτό δεν σα έλεσε τον λόγο. Κυρία Γκέρλιν, έχετε το λόγο. Δύο πράγματα. Πρώτον, η έκθεση εστιάζει αποκλειστικά στις σχέσεις στο πλαίσιο συμφωνιών και θέλω να πω ότι υπάρχουν δύο τομείς εκτός Το ΙΚΑΟ και IMO, δηλαδή Διεθνή Οργάνωση Πολιτική Αεροπορία και Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, που και οι δύο οργανισμοί είναι σημαντικοί. Θα επηρεάσουν αυτού του ε, νέου στόχου. Έχει μείνει εκτό και νομίζω ότι θα έπρεπε ρητά να συμπεριληφθεί. Ο τομέας της ναυσιπλοείας και των αερομεταφορών είναι πολύ σημαντική. Ιδίω η ΔΟΠΑ. Είναι σημαντική για τι αναπτυσσόμενε χώρες, πώ επηρεάζει τις αερομεταφορές και η στάση των αναπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων είναι τελείως διαφορετική. Και αυτό καταδεικνύει σαφέστατα το δίλημα που έχουμε σήμερα. Κάποιες χώρες δηλαδή σηκώνουν πολύ μεγαλύτερο βάρος από κάποιες άλλες. Εδώ στο Κοινοβούλιο τους δύο αυτούς οργανισμούς δεν τους αντιμετωπίζουμε με ικανοποιητικό τρόπο κατά την απόψή μου. Δεν είναι μόνο η ΕΝΒΗ, είναι και η Επιτροπή Μεταφορών και είναι και η ΓΔ MOVE, κάπως περίπλοκα τα πράγματα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δούμε στην έκθεση, γιατί αν θέλουμε να έχουμε αυτή την διπλωματία στον τομέα του κλίματος, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε τους οργανισμούς αυτούς για και με τους οποίους δεν έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη προσέγγιση. Επίσης, η μόχλευση. Το πώς μπορεί να επηρεάσει η υποκρατική διπλωματία με τα, ε, παραδείγματος χάρη με τις ΗΠΑ, τις πολιτείες, τις ξεχωριστές ή επίσης και την Κίνα ως εταίρο απουσία πλέον τον είπα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλους τους άλλους. Μελά. Δύο παρατηρήσεις απλές. Πρώτο, πράγματι, στην έκθεση αυτή τα κράτη μπαίνουν ε, στο 16 και στο 19 σε δευτερεύουσα θέση. Γίνεται λόγο συνέχεια για Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, ενδιαφέρουσα και αυτή η βαθμίδα και αυτή η κλίμακα, αλλά δεν πρέπει να είναι η μόνη. Επίσης, είμαστε επιφυλακτικοί, πάντοτε ήμασταν και θα είμαστε σε σχέση με το πώς μπορεί αυτή η κλιματική αλλαγή να αποτελεί αντικείμενο χειραγώγησης και εκμετάλλευση και οικονομικούς λόγους. Δύο προβλήματα ουσίας υπάρχουν και θέλω να τα αναφέρω. Και η Επιτροπή Περιβάλλοντος και η Επιτροπή Εξωτερικών θα πρέπει να τα έχουν υπόψη τους ότι αυτή τη διπλωματία για το κλίμα. Το πρώτο αφορά την παραγωγή ε, και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας ε, και κάτι που έχουμε καταλήψει εδώ και χρόνια. Να έχουμε πραγματικά συστήματα και πραγματική συνεργασία στον τομέα της άρτευσης, ιδίω για την υποσαχάριο Αφρική. Βλέπουμε να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη συγκέντρωση ε, πολλών στις πόλεις και είναι ένα βασικό θέμα που το έχουμε λίγο πολύ παραγνωρίσει δίνοντας ε, βάρος σε κάποια πιο γενικά κόνσεπτ. Ίσως πρέπει να επανέλθουμε σε αυτά τα βασικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές. Αυτό που έτσι όλοι και εγώ θέλω να το υπογραμμίσω. Και για τον ΙΚΑΟ και για τον ΑΙΜΟ πρέπει να έχουμε αναφορά ξεκάθαρη. Έχω την εντύπωση ότι οι δύο οργανισμοί αυτοί, παρότι είναι που την εγγρατώει, είναι κάπως ε, απομονωμένοι, ε, κάνουν τη δική του ζωή κατά κάποιο τρόπο αλλά συσχετίζονται ε, με αυτά που γίνονται στον ΟΗΕ. Και ήμουν και στην Γενική Συνέλευση. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το τονίσουμε και πρέπει να το συμπεριλάβουμε στους οργανισμούς. Θέλω να πω και κάτι άλλο που θεωρώ σημαντικό για αυτό το σχέδιο έκθεσης των δύο συναδέλφων κυρία Ντάλη εκπροσωπεί βέβαια τον κύριο Λάινεν. Για το σημείο 13 συγκεκριμένα, για τη διεθνή ε, συνθήκη στο μέλλον, ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε μια ρήτρα για τη συνεργασία, για τον τομέα της προστασίας του κλίματος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ. Thank you very much. Anyone else? Uh, Υπάρχει κάποιο άλλο. Αν όχι, εδώ ολοκληρώθηκε ο κατάλληλο των ομιλητών και δίνω ξανά το λόγο ή μάλλον το Προεδρία στον κύριο Μπούχνερ για να ολοκληρώσετε εσεί από πλευρά τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Σα ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε την ε, Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Δράσης. Είναι εδώ εκπρόσωπο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που είμαι εδώ για να σχολιάσω το σχέδιο έκθεσης. Το είπαν πολλοί ότι είναι πολύ επίκαιρη η έκθεση αυτή. Είναι κρίσιμα το 2018 για τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού. Αλλά επίσης κρίσιμο είναι να εκμεταλλευτούμε το παράθυρο ευκαιρίας για να μειώσουμε την υπερθέρμανση στους 2 ή ίσω και τον 1,5 βαθμό Κελσίου. Γιατί προ το παρόν αντιμετωπίζουμε μεγάλε δυσκολίες σε αυτούς τους στόχους. 26 Φεβρουαρίου είχαμε τα συμπεράσματα από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για την Κλιματική Διπλωματία και εκεί παρέχεται μια ξεκάθαρη καθοδήγηση. Και εκεί τίθεται για το θέμα ε, της κλιματικής ανασφάλειας ε, και αναφέρονται και οργανισμοί ε, ΔΟΠΑ και Διεθνής οργανισμοί, Οργανισμός. Πράγματι ζητείται σημαντικό επίπεδο φιλοδοξίας. Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη τις γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές προκλήσεις. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανακτήσουμε την ηγετική μας θέση για να επηρεάσουμε τους άλλους εταίρους και να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία. Έχουμε και το Κατοβίτσι στην Πολωνία που επίκειται. Για την ΕΕ εδώ που εκπροσωπώ. Κάποια στοιχεία. Κλιματική αλλαγή. Είναι στο σταυροδρόμι δύο πολύ βασικών προτεραιοτήτων και στρατηγικών. Πολυμερή, πολυμερή στάση ενίσχυση ασφάλειας και σταθερότητας με την πρόληψη για την αντιμετώπιση των βασικών αιτίων. Μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και έχει και σημαντικό ρόλο η αλλαγή του κλίματος. Υπάρχει αυτή η σχέση εσωτερική και εξωτερική. Το είπατε και ορισμένοι από εσά όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Και αν θέλουμε, μάλλον αν ήμασταν επιτυχημένοι κατά το παρελθόν ιδίω καθόταν προ την cop αλλά και μετά, είναι γιατί ποιος πιέσαμε να υπάρχει έγκαιρη επικύρωση και υλοποίηση και θέση ισχύ τη στο των Παρισίων. Αυτό το κάνουμε γιατί είμαστε αξιόπιστοι. Όχι λόγω της τάσης μας και των δεσμεύσεών μας, αλλά και γιατί συμπεριφορά που που έχουμε και τους στόχους που πετυχάνουμε εσωτερικά και που στηρίζουμε και άλλους να τους πετύχουν. Πολύ σημαντικό το μήνυμα που στέλνουν οι επιτροπές ΕΝΒ και ΑΦΕΤ, συντάσσοντας από κοινού την έκθεση. Έτσι έχουμε τις δύο διαστάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, οι συζητήσεις που θα γίνουν εδώ για το μέλλον του π θα είναι πάρα πολύ σημαντικέ και για αυτέ τι συζητήσει για την κλιματική διπλωματία. Θέλω επίση να πω το εξή. Την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Κομισιόν να εξετάσει θα γίνει μετά τον ορίζοντα το χρονικό του 2030. Μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 19 να έχει παρουσιάσει μια συνολική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Άρα μιλάμε για φιλοδοξία και αξιοπιστία. Εκεί εντάσσονται αυτά. Κάποιες άλλες σύντομες παρατηρήσεις ότι αφορά πάντα την ΕΙΕΔ. The first one indeed is about... Πολυμερές σύστημα πρώτο. Το λέει και έκθεση. Το κλίμα γιατί μας απασχολεί. Το λέει και έκθεση παραλαμβάνω. Γιατί κατά πολέμηση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να προωθήσει την διεθνή συνεργασία. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Δεν μιλάμε μόνο για τη θεματική προσέγγιση εδώ, αλλά για τη διεθνή νομιτάξη και την διεθνή συνεργασία, ιδίω βλέποντα ότι κάποιε χώρε αποσύρονται από αυτή τη συνεργασία. Δεύτερη παρατήρηση. Πολυεπίπεδη διπλωματία είναι η κλιματική διπλωματία. Το είπατε πολλοί από εσά. Ιδίω μετά το Παρίσι, η κλιματική διπλωματία έχει να κάνει με κράτη, μάλλον με κρατικούς φορείς αλλά και με μη κρατικούς φορείς. Είναι παγκόσμια αυτή η δράση. Και οι μη κρατικοί φορείς επίσης πρέπει να συσφέρουν σε αυτήν την υπόθεση. Κάτι εξίσου σημαντικό είναι η πρόθεση του Ευρωκοινοβουλίου και το χαιρετίζουμε αυτό να δώσει μεγαλύτερο ρόλο στην κοινοβουλευτική διπλωματία που είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την δράση στον τομέα του κλίματος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα σημαντικό παίκτη στην πολυεπίπεδη αυτή διπλωματία της Ένωσης και προσβλέπουμε στην ανάπτυξη πρακτικών μεθόδων ανταλλαγής οπότε ε, και συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κλίμα και ασφάλεια. Δεν θέλω να ευσάλθω σε λεπτομέρειες, αλλά είπατε πολλοί από εσάς για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ότι και όπως φαίνεται και από την έκθεσή του βάζει μεγάλη έμφαση στον περιβαλλοντικό και κλιματικό κίνδυνο. Αλλάζει το τοπίο των κινδύνων στην εποχή που ζούμε. Και αυτό είναι ένα θέμα για τη διπλωματία στον τομέα του κλίματος. Και έχουμε και τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Κλιματική διπλωματία αφορά και το 16 για την ειρήνη και την ε, ασφάλεια. Το 16ο στόχο δηλαδή. Καλωσορίζουμε την έκθεση και με τα χαρά να συνεχίσουμε τις συζητήσεις για την κλιματική διπλωματία στο μέλλον. Ευχαριστώ. You very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντελίλ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Έλληνα Μπάτλαρ που εκπροσωπεί την Κομισιόνο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να συζητήσουμε ένα θέμα που θεωρούμε πρωταρχική σημασία για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή στο τομέα της δράσης ε, για το κλίμα. Ε, άκουσα πολύ προσεκτικά τις ε, παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και την ε, υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, εισηγητές, τον κύριο Λίτσκετ τον κύριο Λάιναν και τις ε, επιτροπές για την εξαιρετική δουλειά τους. Το σχέδιο έκθεσης αποτελεί μια πολύ καλή βάση και σημαντική συμβολή για τις μελλοντικές συζητήσεις για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να τονίσω το διαθεσμικό χαρακτήρα της κλιματικής διπλωματίας. Η περσινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη στον τομέα του κλίματος η κυβέρνηση του Τραμπ ανακοίνωσε την αποφασή της ή τουλάχιστον την πρόθεσή της να αποχωρήσει από την Συμφωνία του Παρισιού και ταυτόχρονα είχαμε πάρα πολλά καταστροφικά ε, κλιματικά ε, γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Ήταν ενθαρρυντικό ε, το ότι διαπιστάσουμε ότι παρά την ανακοίνωση του κυρίου Τραμπ, η διεθνή κοινότητα ένωσε τις δυνάμεις της και έδειξε μια μεγάλη αποφασιστικότητα, εξέφρασε ένα όραμα και τη διάθεσή της να ε, προχωρήσει. Σήμερα θα ήθελα να σας πω τρία πράγματα. Το πρώτο αφορά το γενικότερο, το παγκόσμιο πλαίσιο, όπως είπε η συνάδελφος, φετινή χρονιά θα είναι μια δοκιμασία για ε, την ε, αξιοπιστία των ε, συζητήσεων για το κλίμα και των συμφωνιών. Γιατί τρία χρόνια μετά την συμφωνία του Παρισιού, ο κόσμος θα περιμένει να δει πρόοδο. Και φυσικά εδώ έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τους διεθνείς εταίρους μας. Επιπλέον, το πρόγραμμα δράσεων της Συμφωνίας του Παρισιού που θα ε, ορίσει τις λεπτομέρειες της ε, κινητοποίησης και τις διατάξεις που αφορούν τη λογοδοσία των ε, φορέων. Η φιλοδοξία είναι κάτι που θα πρέπει να έχει και πρακτικές διαστάσεις. Ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλές συζητήσεις στα πλαίσια του ε, πλαισίου για την ε, ενέργεια και το κλίμα και φαίνεται ότι υπάρχει η βούληση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο. Υπάρχουν ε, γενικές πολιτικές και μέτρα και πρέπει να ε, συνεργαστούμε με τους εταίρους μας προκειμένου να διασφαλίσουμε μια μετάβαση προς μια οικονομία με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και να δημιουργηθούν ανοίγματα προκειμένου να μοιραστούμε την εμπειρία μας και να προωθήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα για την ενίσχυση των συνεργασιών και με τις αναπτυσσόμενες ε, οικονομίες οι οποίες ε, αντιπροσωπούν ε, σημαντικό κομμάτι των εκπομπών άνθρακα. Πέρα από τις στρατηγικές συνεργασίες με τις μεγαλύτερες οικονομίες, πρέπει να επιδείξουμε και αλληλεγγύηση και πέρα από τις χρημα χρηματοδοτήσεις ε, θα πρέπει να ε, δράσουμε, η δραστηριοποίησή μας θα είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να οικοδομήσουμε συνεργασίες και συμμαχίες προκειμένου να διασφαλίσουμε τις απαραίτητες δράσεις για την, ε, να ολοκληρωθεί το rulebook του Παρισιού. Το τρίτο που θα ήθελα να πω είναι γιατί αυτή η έκθεση είναι ιδιαίτερα επίκαιρη. Όπως είπατε πολλοί από εσά, αυτή τη στιγμή συζητάτε το επόμενο πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε το στόχο του 20% ε, χρηματοδότηση στο επόμενο πλαίσιο. Θα ήταν περίεργο αν δεν ε, ε, στοχεύαμε ένα υψηλότερο στόχο στο μέλλον. Η έκθεση αυτή και ο επίκαιρος χαρακτήρας της ε, σχετίζεται και με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει μεγάλη σημασία για τους Ευρωπαίους πολίτες. Πρόκειται για σημαντικό ορόσημο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να βασιστούμε στις ε, δυνάμεις μας και στα ε, πλεονεκτήματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Τέλος, αυτή η έκθεση είναι πολύ επίκαιρη γιατί υπογραμμίζει την σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στους κρατικούς φορείς, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, δεσμούς και στα πλαίσια του Διεθνούς Προγράμματος Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να ε, το δουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Είναι σημαντικό να υπάρχει ε, ενότητα ανάμεσα στους διάφορους ε, φορείς, συνεργασία και είναι σημαντικό να εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα φιλόδοξο όραμα και κάλεσε την Κομισιόν να υποβάλει την ενδιάμεση στρατηγική της η οποία είναι προτερική σημασία σε αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λίτς, θέλετε να εκφράσετε κάποια συμπεράσματα. Ναι, ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους ε, συναδέλφους από την Κομισιόν και ε, που υπογραμμίσετε κάποια θέματα και προσθέσατε και καινούρια. Θα εξετάσω επιμέλως τις ε, προτάσεις αυτές. Ε, περιμένω και τις τροπολογίες. Φαίνεται ότι το θέμα αυτό είναι πολύπλοκο. Έρχεται καλοκαίρι και θα ήθελα να τονίσω διάφορα θέματα που εκφράσατε ε, και εσείς όλα τα θέματα καλύπτονται από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και πρέπει να τους λάβουμε υπόψη. Μιλήσατε για την ε, επιστημιστική ασφάλεια, το, την ποιότητα του νερού, το, τη σημασία του πόσιμου νερού. Το θέμα των εμπορικών συμφωνιών αναφέρθηκε πολλές φορές. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, μιας και με τη συμφωνία ΣΥΤΑ με το Καναδά έχει ξεκινήσει η υλοποίηση και θα πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, πολλά ζητήματα σχετικά με τη φτώχεια φτώχεια και τις κοινωνικές διαστάσεις και το ρόλο τους σε αυτό το τομέα. Τέλος, αναφέρθηκε το θέμα της, ε, των δράσεων για το κλίμα των ε, εταίρων μας. Είναι σημαντικό να ε, υπάρξει συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αντιπροσωπείες όχι μόνο των δικών μας επιτροπών, προκειμένου όλες οι επιτροπές να έχουν μια επαφή με τις συνεργαζόμενες ε, χώρες, προκειμένου να συλλέξουμε πληροφορίες, να ε, έχουμε αποστολές επιτόπου και είναι σημαντικό να ε, ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Μετά ε, ενωμένω και τις επόμενες ε, συνεδριάς σχετικά με αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λίτς. Η παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης τονίζει τη σημασία ε, αυτού του θέματος στο πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, τους εισηγητές, τους και όδους εισηγητές, τους συμμετέχοντες και φυσικά τους εκπροσώπους της Κομισιόν και της ε, ΕΙΕΔ. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και για το γεγονός ότι τονίζετε το σημαντικό ρόλο της κλιματικής διπλωματίας και για την ε, σημασία της συνεκτικής δράσης για το κλίμα και τη στήριξη των θεσμεύσεων στα πλαίσια της Συμφωνίας του ε, Παρισιού, στα πλαίσια του προγράμματος δράσης μέχρι το 2030. Ευχαριστώ τους. Ε, ε, ε, αναμένω και τις συζητήσεις, τις μελλοντικές σχετικά με αυτό το πολύ σημαντικό θέμα τις ερχόμενες εβδομάδες. Ποιες είναι οι προθεσμίες, οι καταληκτικές ημερομηνίες για την κατάθεση των τροπολογιών 11 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι, στις 16 Μαΐου θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση και τον Ιούλιο του 2018 θα γίνει ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και την παρουσία σας εδώ.